Καλή σας μέρα. Καθίστε παρακαλώ. Έχουμε ψηφοφορίες. Χρειάζεστε την ε, κάρτα σας για ηλεκτρονική ψηφοφορία. Καθίστε. Ready? Okay. Thank you very much. Έτοιμοι? Ωραία. Να συγκεντρωθούμε. Πρώτα θα ψηφίσουμε προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο σχετικά με τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στη Βόνη. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. And the vote is closed. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στην προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή για το ίδιο θέμα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο απόφασης του Σεβουλίου για την τροποποίηση του Κιγκάλι στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφονται στη βάδα του Όζοντος. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά πάντα. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Ψηφίζουμε τώρα το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την αποδοχή της τροποποίησης το πρωτόκολλο για την ε, ρήπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση και μείωση όξης ευστροφισμού και τρυποσφαιρικού όζοντος. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Τώρα φτάνουμε στην αντίρρηση, ένσταση σχετικά με την απαγόρευση της δραστικής ουσίας της θιαμοξίνης. Παρακαλώ, ψηφίστε ηλεκτρονικά. Θιαμοθοξάμι. Λήξη της ψηφοφορίας απορρίφθηκε. Τώρα ψηφίζουμε την ε, ένσταση σχετικά με την έγκριση της δραστικής ουσίας ημιντακλοπρίτ. Ψηφίστε παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Ένσταση τώρα για την έγκριση της δραστικής ουσίας κλωθιανιδένης. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τώρα ψηφίζουμε για την φαλαινοθυρία στην Νορβηγία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Αυτές ήταν οι σύντομες ψηφοφορίες και τώρα περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Πρόκειται για τη στόχους βιωσιμότητας. Έκθεση DANS, δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της βιωσιμότητας. Είσαστε έτοιμοι? Ωραία. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Φαρία απέσυρε την τροπολογία του 290. Συμβαστική τροπολογία 1 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεβε 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 55 Καταπίπτει όμω. Συμβαστική 36 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 71 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 71. Ψεφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές. Θα λέξουμε για τη συμβαστική 7. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρες τη ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Τροπολογία 73 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 79 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 97 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 99 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 107 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 108 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 110 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 112 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 129 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 31 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ωραία, θα ελέγξουμε για τη σεβαστική 31. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, ψηφίστε. Πέρας της φοφορίες. Απορρίφθηκε. Αλλά εντάξει, ισοψηφία. Ναι. Συνεπώς πρέπει να ψηφίσουμε για τις τροπολογίες που καλύπτονταν. 130 πρώτα πέρ. κατά, αποχές. Θα λέξουμε; γιατί δεν είδα χέρια να σηκώνονται. 130 λοιπόν, ηλεκτρονικά ψηφίστε. Πέρα στις φοφορίες. Εγκρίνεται. Άγκρι 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Αλλά ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις φοφορίες. Εγκρίνεται, ναι. Άγκρι 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άγκρι 9, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 14, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 135, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 142 υπέρ. Α, πρόκειται και για κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω, να σε ελέγξουμε για την 145. Ψηφίστε. Πέρα τις Εγκρίθηκε. 146 δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 148 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 149 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. 149 ηλεκτρονικά, ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε. 150 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 151 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 155 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 163 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 165 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 166 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 170 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεβε 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 178 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ωραία, για την 178 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της φοφορίας. Συγγνώμη. Έκανα λάθος, λέει πρόεδρος, όντως εγκρίνεται. 179 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 180 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 182. Α, και η 181, γιατί δεν ε, πέρασε ο συμβασμός, υπέρ παρακαλώ της 181, κατά, αποχές, απορρίπτεται νομίζω, αλλά ελέγξουμε. 181. Είναι τσίμα τσίμα και αλλάζουν οι πλειοψηφίες. Να, εγκρίθηκε. 182 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 183 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 177 υπέρ, κατά, Αποχές. Θα ελέγξουμε. 177. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. <clears throat> Πέρα στις ψηφοφορίες. Και εγκρίθηκε. 185 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. 186. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. <clears throat> Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Συμβαστική 16 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Κάποια παρέμβαση εκτός μικροφώνου, δεν την ακούμε. δεν ακούγονται αγγλικά γιατί μιλάω αγγλικά, λέει. Γιατί φαίνεται διαμαρτυρήθηκε για την αγγλική διερμηνία η ομιλήτρια, αλλά αφού μιλάει αγγλικά η πρόεδρο, δεν υπάρχει αγγλική διερμηνία. Εντάξει τώρα. Ωραία, θα προσπαθήσω να μιλάω πιο κοντά στο μικρόφωνο. Συμβαστική 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καλτ 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεβε 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεβε 7 υπέρ, α όχι, καταπίπτει, καταπίπτει. Δεβε 15 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 20 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, Πρώτο τμήμα πάλι υπέρ, εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 203. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 204. Καταπίπτει. 205. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2.15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 216 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 217 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 223 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 224 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 226 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Αν Α, θέλετε να ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά 226. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 230 υπέρ. Κατά. Αποχές Αγκρίνεται. 231 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 232 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα έχουμε τροπολογίες Επιτροπής Πολιτισμού. Και αρχίζουμε από την 11 υπέρ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 κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, τροπολογία 237 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 238 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 239 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 240 υπέρ, κατά, αποχές θα ελέγξουμε. 240 ελέγχουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας τις ψηφοφορίες. εγκρίθηκε. 241 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 246 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 248 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 253 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 254 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 259 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 260 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε. 260. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε. 262 τώρα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 263 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 264 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 265 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε για το δεύτερο τμήμα. Ηλεκτρονικά ψηφίστε παρακαλώ. εγκρίθηκε. ΔΕΒΕ 18 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την ΔΕΒΕ 18. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 271 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε. 271 για το πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της φοφορίας. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 272 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 274 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 277 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 278 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 280 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 281 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 282 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 283 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 30 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε για την συμβαστική 30. Συμφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. πέρασε της Εγκρίθηκε. Τώρα έχουμε μία σειρά από τροπολογίες της Επιτροπής Γεωργίας, Αγκρή. Θα λέω τα νούμερα μόνο, έτσι. Αγκρή 6. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Πιστεύω, αλλά ας ελέγξουμε για την 20. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρες της φοφορίας. Εγκρίθηκε. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε για την 22. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρα στις φοφορίες. Και εγκρίθηκε. Δεν σηκώνετε τα χέρια σας όμως. Γι' αυτό χρειάζεται να κάνουμε ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Θα το είχα δει. Άγκρι 23 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 295 τώρα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Καλτ 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 296 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 299 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 300 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αναλέξουμε. Ωραία. Γιατί είναι 300. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Α, απορρίφθηκε. Εντάξει. Ναι. Δεν είχα καταλάβει τι λέγατε. Πέρα στις ψηφοφορίες, ναι, προφανώς απορρίφθηκε. 302 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε. 302. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε. ΔΕΒΕ 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 305. Υπέρ. Ή όχι. Όχι, δεν ψηφίζουμε για 305. 308 τότε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία αριθμός 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 3 και 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 32 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12 ή όχι. Όχι. Συμβιβαστική 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύε Αλφα. υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεβε β υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεβε σ γάμα υπέρ, κατά, αποχές θα ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 35 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε τροπολογία 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30... Τριάντα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύε διάφορες τροπολογίες. Η πρώτη είναι η D, δέλτα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η ε υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε για την ε. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας, εγκρίνεται. F, σίγμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. G, ζήτα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και H, ήτα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τώρα, τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίθηκε. Τελείωσαν οι ψηφοφορίες λοιπόν εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Συνάδελφοι, να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα γιατί έχουμε προχωρήσει λίγο πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε, οπότε θα συνεχίσουμε στις 10. Έχετε λίγο καιρό για να πιείτε έναν καφέ.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 Well, hello. Um, next item on our agenda is the exchange of views with the Commission on refit of Περνάμε στο επόμενο σημείο, δηλαδή αξιολόγηση ρηφή ε, της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων. Ε, και έχουμε και τους ε, προσώπους της Επιτροπής, ο κ. Πάκο νομίζω είναι μαζί μας, επικεφαλής της ε, μονάδας ε, της, ε, σχετικής μονάδας της Γενικής Διευθύντης Κλίματος. Θεωρούμε λοιπόν το ρήφι σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό ακριβώς σας ζητήσαμε να προσέλθετε σήμερα εδώ και να μας κάνετε μια παρουσίαση του γράφου εργασίας της Επιτροπής. Οπότε θα μας κάνετε την παρουσίαση. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε σήμερα εδώ να σας ε, παρουσιάσουμε αυτή την αξιολόγηση της ε, οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων. Όπως γνωρίζετε η εν λόγω αξιολόγηση δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο του πακέτου για την κινητικότητα που υιοθετήθηκε τον περσινό Μάιο. Και θα ήθελα να σας κάνω μια γενική επισκόπηση ε, της ε, οδηγίας ε, προτού προβώ στα πορίσματα της αξιολόγησης. Η οδηγία λοιπόν για την ποιότητα των καυσίμων είναι σχετικά παλαιά. Υιοθετήθηκε δηλαδή σχεδόν πριν από 20 έτη και έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα. Όμως οι κύριοι στόχοι της παρέμειναν οι ίδιοι. Και όπως βλέπετε εδώ στην διαφάνεια είναι η επίτευξη υψηλού επίπεδου προστασίας ε, του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, βελτίωση της ε, ποιότητας ε, της ατμόσφαιρας, βελτίωση της λειτουργίας της οδικής μεταφορέ για τα καύσιμα και για τα οχήματα και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Και προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η μείωση των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών, θα πρέπει κανεί να εξετάσει όλους, ε, όλα τα συστατικά, αν θέλετε, στοιχεία των μεταφορών και σε αυτά συγκαταλέγονται τα καύσιμα, δηλαδή η μείωση των εκπομπών άνθρακα από τα καύσιμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία τη αξιολόγηση, ε, να πούμε ότι ε, βασίστηκε σε μια εξωτερική μελέτη, την οποία ανατέθηκε από την Επιτροπή και η οποία έχει υιοθετηθεί στην βιβλιοθήκη στο Bookshop της επιτροπή και επίσης ε, η λόγω μελέτη ή μάλλον η αξιολόγηση έλαβε χώρα σε στενή συνεργασία με εμπλεκόμενου φορεί, με κυβερνητικέ οργανώσει, κράτη-μέλη ε, και ε, οργανώθηκε και ένα workshop στο οποίο αναδείχθηκε μια ευρεία συνένεση ως προς τα ζητήματα που εξέτασε η αξιολόγηση. Εκείνο που θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω είναι το εύρος της παρούσας αξιολόγηση. Η αξιολόγηση λοιπόν δεν καλύπτει το σύνολο των διατάξεων της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων αλλά δύο εξαιρεσει υπάρχουν, δύο διατάξεις οι οποίες δεν καλύφθηκαν. Ε, ε, μία από αυτές είναι ο στόχος ε, της μείωσης των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, αυτό το άρθρο 7α, που θέτει τον στόχο της μείωσης αυτών των εκπομπών κατά 6% στο 2020 και δεν περιλήθηκε σε αυτή την αξιολόγηση, σε αυτή τη διάταξη, γιατί ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη. Οπότε όταν κανείς αξιολογεί κάτι θα πρέπει να κάνει μια ανασκόπηση ε, του πώς έχει πραγματοποιηθεί η ε, υλοποίηση, η εφαρμογή στην πράξη της εν λόγω διάταξης. Αφού λοιπόν αυτό το τμήμα της ε, ε νομοθεσίας μεταφέρεται τώρα στην Εθνική Νομοθεσία και η προθεσμία για τη μεταφορά ήταν ε, ο Απρίλιος τώρα φέτος, η αξιολόγηση θα εξηγήσει από εδώ και στο εξή. Η δεύτερη διάταξη που εξαιρέθηκε από την αξιολόγηση είναι τα κριτήρια για την βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων, που ε, ε, έχει ήδη αξιολογηθεί στο παρελθόν. Άρα, προτού περάσω στα συμπεράσματα της εν λόγω αξιολόγησης, θα ήθελα να σας πω δύο λόγια ε, σε σχέση με τις κύριες διατάξεις αυτής της οδηγίας. Το πιο σημαντικό είναι ότι ε, προβλέπει συγκεκριμένες ε, προδιαγραφές σε ό,τι αφορά τη βενζίνη, ε, το πετρέλαιο και τα συστατικά τους και ο κύριος στόχος είναι η μείωση των ατμοσφαιρικών ρήπων. Και εδώ στην διαφάνεια βλέπετε τους κύριους ατμοσφαιρικούς ρήπους οι οποίοι ακριβώς εμπίπτουν στις διατάξεις των προδιαγραφικών καυσίμων της οδηγίας. Δηλαδή βλέπουμε εδώ οξύδια του θείου, εκπομπές ειδικότερα μολύβδου, ε, σωματίδια και κάποιους ε, υδρογονάνθρακες. Επίσης, ε, Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογή αυτή τη οδηγία. Αφορά στα καύσιμα τα οποία χρησιμοποιούνται στι οδικέ μεταφορέ και υπάρχουν και ε, κάποιε πλέον προδιαγραφέ, αλλά πιο, όχι τόσο αυστηρές σε ό,τι αφορά τα ε, μη οδικά κινητά μηχανήματα. Ε, πέραν αυτών των διατάξεων ε, θα πρέπει να έχουμε κατά νου η εν λόγω οδηγία θέτει κάποια όρια σε ό,τι αφορά την τάση ατμών για ορισμένα είδη βενζίνες προκειμένου να αποφευθεί η διαφυγή εξατμίσεων για παράδειγμα στο πλαίσιο της ή από τη δεξαμενή καυσίμου ή κατά την λειτουργία ανεφοδιασμού με καύσιμο. Επίσης ο στόχος, οι διατάξεις στοχεύουν στο να υπάρχει να είναι να είναι συμβατά αυτά τα καύσιμα με, τις, ε, με τους νέους κινητήρες και την ε, επεξεργασία των ε, καυσαρίων τους. Δηλαδή, το σημαντικό είναι, ένα σημαντικό στόχος είναι όταν γίνεται ανεφοδιασμός με το συγκεκριμένο καύσιμο του οχήματο να μην δημιουργείται ζημία στο κινητήρα του καυσίμου. Και γι' αυτό ακριβώς έχουν τεθεί συγκεκριμένα όρια ανάμειξη συγκεκριμένων βιοκαυσίμων καθώς αυτά δεν είναι συμβατά με όλα τα είδη κινητήρων. Τα δύο κύρια όρια λοιπόν μειγμάτων ε, που αναφέρονται σε αυτή την οδηγία είναι ε, το περιεχόμενο ε, σε βιοκαύσιμα των καυσίμων που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 7% και μετά η εθανόλη η οποία στην βενζίνη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 10%. Ε, Αυτά λοιπόν τα ε, δύο όρια έχουν τεθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των κινητήρων που τα λόγω καύσιμα. Όμω υπάρχουν και κάποιε παρεκκλήσει οι οποίε ε, μπορούν να εφαρμοστούν ειδικότερα σε ό,τι αφορά το βιοντίζελ και σε ό,τι αφορά και την, τα όρια τάση ατμών. Κάτι ακόμα που είναι σημαντικό σε αυτή την οδηγία είναι ότι υπάρχουν ε, ε, ότι υπάρχει ένα πολύ αυστηρό σύστημα παρακολούθησης ποιότητας των καυσίμων, το οποίο θα πρέπει να δημιουργήσουν τα κράτη-μέλη. Οπότε υπάρχει, έχει δημιουργηθεί δηλαδή ένας καλός μηχανισμός υποβολή αναφορών προκειμένου η Επιτροπή να μπορεί να αξιολογεί τη συμμόρφωση με τι διατάξει τη οδηγία. Υπάρχουν ετήσιε εκθέσει οι οποίε υποβάλλονται και δημοσιεύονται ετησίω από την Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντο, τον EEA. ΕΕ. Ας περάσουμε τώρα λοιπόν στα ε, απορίσματα αυτής της αξιολόγησης και θα δούμε εδώ τα κύρια κριτήρια, το οποίο γνωρίζετε, καταρχήν η αποτελεσματικότητα ε, της ε, νομοθεσίας αυτής της οδηγίας. Εδώ βλέπετε λοιπόν σε αυτά τα γραφήματα ποια είναι η εξέλιξη σε ό,τι αφορά τους κύριους ρήπου από το 1995 και μετά στο, ε, καθ' όλη τη διάρκεια της ε, εφαρμογής λοιπόν αυτής της οδηγίας διαπιστώνουμε ότι όλοι οι κύριοι ατμοσφαιρικοί ρήποι μειώθηκαν σε σημαντικό βαθμό και αυτό αποτέλεσε σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα των προδιαγραφών σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, ειδικότερα τα όρια σε σχέση με το θείο, ε, το μόλιδο. Αυτά λοιπόν τα όρια που τέθηκαν μέσω της οδηγίας είχαν άμεσο και σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση των σχετικών εκπομπών. Όμως ε, δεν ήταν αυτός ο μόνος λόγος γιατί και τα πρότυπα που ορίστηκαν για τις ε, εκπομπές ε, των οχημάτων ε, συνέβαλαν. Δηλαδή τα πρότυπα αυτά ήταν δυνατό να εφαρμοστούν μόνο εφόσον είχε βελτιωθεί η ποιότητα του καυσίμου. Δηλαδή όταν είχαμε καύσιμο υψηλή περιεκτικότητα σε θείο δεν επέτρεπε το ενόγο καύσιμα, καύσιμο ο καταλήτης του αυτοκινήτου να λειτουργήσει σωστά. Άρα λοιπόν τα, οι προδιαγραφές που θέσαμε σε ό,τι αφορά τα καύσιμα και οι προδιαγραφές που θέσαμε σε ό,τι αφορά τους συνετήρες των καυσίμων οδήγησαν συνδυαστικά στους μειώσει των κύριων ατμοσφαιρικών ρήπων που παρατηρούμε εδώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά και πάλι την αποτελεσματικότητα, εξετάσαμε και τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ε, των καυσίμων. Εδώ λοιπόν το πόρισμα μας είναι θετικό, δηλαδή στο 99 έως 100% των περιπτώσεων έχουμε πλήρη συμμόρφωση, οπότε ε, θεωρούμε πως ναι εφαρμόζεται πολύ σωστά ε, παρούσα οδηγία. Επίση, στο πλαίσιο τη διαβούλευση που έγινε με του ενδιαφερόμενου φορεί, ε, διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχαν ενδείξει ότι έχει προκληθεί ζημιά στον κινητήρα ή σε άλλα ε, μέρη του οχήματο λόγω ακριβώ χαμηλή ποιότητα του χρησιμοποιούμενου καυσίμου. Άρα λοιπόν αυτό δείχνει ότι το σύστημα παρακολούθηση τη ποιότητα καυσίμου που έχει ακριβώ έδρα, έχει θεσπιστεί από τα κράτη-μέλη, λειτουργεί καλά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κριτήρια που εξετάσαμε, ε, να πούμε ότι ε, δεν ήταν ε, δυνατό να προβούμε σε μια πλήρη αξιολόγηση τη σχέση κόστου αποτελέσματο τη εν λόγω οδηγία. Όμω τα δεδομένα τα οποία έχουμε συλλέξει σε ό,τι αφορά ε, τι δαπάνε για του προμηθευτέ καυσίμου αλλά και για τι εγκαταστάσει τη και των ε, τα συστήματα παρακολούθησης διαπιστώνουμε ότι ε, όλες αυτές οι δαπάνες σίγουρα ε, δικαιολογούνται και υπερτερούνται από την αποφευχθήσα ζημία στο περιβάλλον και στην ανθρώπινα υγεία. Επίσης, με βάση τα ελάχιστα πρότυπα καυσίμου που έχουμε θεσπίσει, οι προμηθευτές καυσίμου ουσιαστικά μπορούν να αναμένουν χαμηλότερες, ε, χαμηλότερα, χαμηλότερες δαπάνες σε σύγκριση με κάποια πρότυπα που θα είχαν θεσπιστεί ανά κάθε κράτος μέλος. Όμως από εκεί και μετά υπάρχει και η ποικιλία των διαφορετικών βιοκαυσίμων. Η οδηγία δηλαδή θέτει κάποιες ελάχιστες ε, απαιτήσει και οι μεγαλύτερες λοιπόν διαφοροποιήσεις που βλέπουμε μεταξύ των διαφορετικών αγορών, εθνικών αγορών καυσίμων είναι ε, διαφορετικές προτιμήσεις σε ό,τι αφορά την ανάμειξη των βιοκαυσίμων. Δηλαδή, στα διάφορα κράτη-μέλη βλέπουμε ότι υπάρχουν και διαφορετικές ε, νομικές διατάξεις ως προς το πώς μπορούν να αναμειγνύονται τα βιοκαύσιμα σε κανονικά καύσιμα. Και αναφέρθηκε λοιπόν στο πλαίσιο τη διαβούλευση ότι θα μπορούσαν να αποφευθούν κάποια κόστη αν ακριβώ αυτή η διαφοροποίηση στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την ανάμειξη των βιοκαυσίμων θα μπορούσε να μειωθεί. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, συνοχή, τη συμμόρφωση δηλαδή με άλλες ε, νομοθεσίες, να πούμε πω εξετάσαμε διάφορε σχέσει, αλλά ένα κύριο δεσμό, μια κύριε σύνδεση αυτή τη οδηγία είναι με την οδηγία ε, ε, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, και όπου έχει τεθεί ο στόχος για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών έως το 2020. Εξετάσαμε λοιπόν πως την, την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων και διαπιστώσαμε ότι ναι, συμμορφούνται με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, στο πλαίσιο πάντα της συνοχής και την εσωτερική συνοχή, διαπιστώνουμε ότι διατάξεις τόσο στο επίπεδο των παρεκκλήσεων όσο και σε ό,τι αφορά τους περιορισμούς εντάσσεται στο πνεύμα της οδηγίας. Ε, ε δηλαδή, ε, λάβαμε υπόψη μας το γεγονός ακριβώς ότι υπάρχουν τέτοιου είδους παρεκκλήσεις και ότι υπάρχουν κάποια είδη καυσίμων τα οποία έχουν εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Άρα λοιπόν, περνώντα στα συμπεράσματα, κυρία Πρόεδρε, ε, να πούμε ότι αυτό που μπορούμε να σας δηλώσουμε είναι ότι η οδηγία για την ποιότητα του καυσίμου είναι κατάλληλη για την προβλεπόμενη χρήση τη, προσθέτει προστιθέμενη αξία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να συνεχίσει να ισχύει γιατί παρέχει ένα υψηλό βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Ε, δεν υπάρχουν ε, ενδείξεις ότι η ευελιξία που έχει προβλεφθεί, δηλαδή τα περιθώρια που έχουν δεθεί για διαφορετικά επίπεδα ανάμειξης βιοκαυσίμων ή οι θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την επίτευξη των βασικών στόχων της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων ή θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποδιοργανώσεις της αγοράς. Άρα λοιπόν ε, φρονούμε ότι σε αυτή τη φάση δεν θα πρέπει να εξεταστεί ε, το ενδεχόμενο αναθεώρησης της οδηγίας για την ποιότητα του καυσίμου. Παρ' αυτά, καθώς η εν λόγω οδηγία δεν έχει ως στόχο την πλήρη εναρμόνιση ε, της ε, ευρωπαϊκής αγοράς ε, μεταφορών και καυσίμων μεταφορών, εμένουμε μόνο σε αυτά τα συμπεράσματα, σε αυτό το επίπεδο. Αυτά από την πλευρά μας. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Um, uh, Ευχαριστούμε πολύ και τον ε, εκπρόσωπο της Κομισιόν για όλα αυτά που μας είπατε. Έχω να κάνω κάποιες ερωτήσεις με βάση αυτά που ακούσαμε και ε, επίσης ε, με βάση αυτά που είπατε κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής απόψεων. Αν κατάλαβα καλά από την ομιλία σας, η οδηγία Ρουφίτ εστιάζει στα πάντα εκτός από το 7α και 7β έως 7η. Το 7α ε, άρχισε να εφαρμόζεται πρόσφατα. Το 7B και 7E αυτή τη στιγμή είναι υπό αξιολόγηση και αναθεώρηση. Και αν ισχύει αυτό, τότε πότε θα έχετε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, κυρίως όσον αφορά τα άρθρα 7, B και E. Και ρωτώ επίσης κατά πόσο η Κομισιόν προτίθεται αργότερα να εφαρμόσει το REFIT και σε σχέση με το άρθρο 7α. Πότε προβλέπετε να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η μία μου ερώτηση. Η άλλη αφορά στο γεγονός ότι παρότι η οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων ε, θεωρεί ότι πρέπει να είναι αποτελεσματική για να υπάρχει υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, εγώ από ό,τι κατάλαβα η μείωση των εκπομπών πολλών ρήπων ήταν πολύ πιο χαμηλή από ό,τι είχε προβλεφτεί. Εσείς το επιβεβαιώνετε αυτό. Και αν ναι, μπορείτε να μας πείτε ποιοι είναι οι λόγοι που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς εξηγεί αυτό το ότι τελικά η μείωση των εκπομπών είναι πολύ πιο περιορισμένη από ό,τι είχε προβλεφθεί αρχικά και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ε, για να υπάρχουν τα ίδια αποτελέσματα που είχαν τεθεί εξ αρχής. Κατά τα άλλα, κάποια στιγμή στην ομιλία σας είπατε ότι τα περισσότερα καύσιμα στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχουν εναρμονιστεί με την οδηγία. Εγώ όμως γνωρίζω νομίζω ότι υπάρχουν κάποια καύσιμα για τα οποία δεν ισχύει αυτό. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλω να ρωτήσω, έχει πληροφόρηση για αυτά τα καύσιμα. Ε, και αυτά τα καύσιμα αφορούν συγκεκριμένα κράτη-μέλη ή αφορούν το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θα ήθελα να εστιάσω και πάλι ε, στο άρθρο 7α, που ξέρω ότι δεν εντάσσεται μέσα στο refit, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον κυρίως για μένα, διότι το άρθρο 7α εστιάζει στη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου ε, κοιτάζοντας βέβαια την ποιότητα των καυσίμων. Και εξ όσων γνωρίζω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτή την προσέγγιση ε, των εκπομπών θερμοκηπίου ε, στην οδηγία περνάει σε μια άλλη προσέγγιση, στην προσέγγιση του όγκου και της ποσότητας. Και θέλω να γνωρίζω κατά πόσον πράγματι αυτό ισχύει, αυτό που λέω, και αν ισχύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι σκέπτεται να κάνει. Και η τελευταία μου ερώτηση είναι η εξής. Ασκείται κριτική προς αυτήν την οδηγία και η κριτική λέει ότι ε, η οδηγία νοθεύτηκε σε μεγάλο βαθμό ε, γιατί ασκήθηκε πίεση από ομάδες και από ε, βιομηχανικούς κύκλους. Εάν λοιπόν αυτό ισχύει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει αυτά τα παραθυράκια, τα κενά, τα χαρακτηρίσουμε και πώς ε, σκέπτεται να ε, ενδεχομένως να τα εντοπίσει και να τα καλύψει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, ερωτήσεις παρακαλώ. Αν όχι, θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Μήπως μπορείτε να μας εξηγήσετε καλύτερα τα στοιχεία που μας παρουσιάσατε, τα γραφήματα που απεικονίζουν τους ρήπους. Μήπως μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς ακριβώς ερμηνεύονται. Γιατί στα γραφήματα βλέπω να υπάρχουν κάποιες ε, κινήσεις ε, σε κάποιους ρήπους, αλλά πάλι σε κάποιους άλλους καμία μετακίνηση. Ίσως μπορείτε λιγάκι να μας το εξηγήσετε αυτό. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος επιθυμεί να υποβάλει κάποια ερώτηση. Αν όχι, θα ήθελα να δώσω ε, και πάλι το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για τις ε, ερωτήσεις. Ε, αν δούμε λιγάκι την ε, αξιολόγηση των τμήματων εκείνων που δεν καλύπτονται από την τρέχουσα αξιολόγηση, ε, σας είπαμε το άρθρο 7α τώρα πλέον εφαρμόζεται. Άρα δηλαδή η αξιολόγηση θα λάβει χώρα μετά την πλήρη εφαρμογή αυτού του άρθρου που ε, ολοκληρώνεται το 2020. Όσον αφορά τα άρθρα 7b και 7e για τα κριτήρια της ε, βιωσιμότητας σε σχέση με τα καύσιμα, η αξιολόγηση έχει ήδη λάβει χώρα και αποτελεί ένα τμήμα της πρότασης για τη νέα οδηγία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεκέμβριο του περασμένου έτους. Εκεί λοιπόν εντάσσεται αυτή η, αυτό το άρθρο. Όσον αφορά τώρα στους ε, ατμοσφαιρικούς ρήπους, και πώς ακριβώς έχουν περιοριστεί σε σχέση με αυτό που αναμενόταν. Αν δούμε λιγάκι την αρχική μελέτη αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τότε που προετοίμαζε την οδηγία, για την οποία μιλάμε σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κάνει κάποιες προβλέψεις ε, και κατέληγε στο ότι θα υπάρξει περαιτέρω μείωση των ατμοσφαιρικών ρήπων. Αλλά δεν συνέβη. Γιατί πρώτον ο όγκος των μεταφορών από τότε που ολοκληρώθηκε η μελέτη αντικτύπου και δεύτερον γνωρίζουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια ανοιχτά θέματα ε, σε σχέση με την ε, ε, μεταχείριση κάποιων καυσίμων και κυρίως όσον αφορά ε, νέες διατάξεις RDE για τα οξύδια του αζότου. Τα καύσιμα, τα οποία δεν συμβαδίζουν με την οδηγία, ε, υπάρχουν παραδείγματα καυσίμων που πράγματι ε, δεν συμβαδίζουν με την οδηγία, δεν ε, σέβονται αυτά τα οποία αναφέρει η οδηγία. Και θα δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου, Όσον αφορά τώρα στο τι θα συμβεί ε, με το θέμα της αφαίρεσης του άνθρακα από τα καύσιμα και κατά πόσον θα πάμε περισσότερο σε μια προσέγγιση όγκου και όχι τόσο ενέργειας κατά το 2030. Ε, η Κομισιόν το Δεκέμβρη του προηγούμενου έτους ε, κατέθεσε μια οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η πρόταση αυτή που στηρίζεται και με μελέτη αντικτύπου. Προτείνουμε λοιπόν να υπάρχει μείγμα υποχρεωτικά για καύσιμα που εκπέμπουν, που έχουν εκπομπές και το κρίσιμο σημείο θα είναι ε, πώς ακριβώς θα συντίθεται αυτό το ενεργειακό μείγμα. Εξάλλου, έγιναν πολλές συζητήσεις ανάμεσα στους νομοθέτες ε, τα τελευταία χρόνια σχετικά με την νομοθεσία. Η νομοθεσία εφαρμόζεται. Βεβαίω, ε, εμεί ε, θέλουμε να αποδοθεί ιδιαίτερη σημασία στα θέματα του ελέγχου και αναφορών περί νομοθεσία για να μπορούμε να αξιολογήσουμε τον όγκο των ε, διαφόρων καυσίμων που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν έχετε να μου υποβάλλετε κάποια συγκεκριμένη άλλη ερώτηση. Απλά ε, θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι όσον αφορά τις εκθέσεις ε, περί τον έλεγχο της ποιότητας, εκεί διαπιστώνουμε ότι σε μεγάλο βαθμό τα καύσιμα έχουν συμμορφωθεί. Ε, δηλαδή η οδηγία ισχύει, τα καύσιμα έχουν προσαρμοστεί κατά 99% όσον αφορά το πετρέλαιο και κατά 100% ε, η βενζίνη δίζελ. Υπάρχουν βέβαια κάποια που δεν καλύπτονται από την οδηγία, αλλά για αυτά τα καύσιμα δεν υπάρχουν και ιδιαίτερε προδιαγραφέ. Αυτό ισχύει κυρίω για καύσιμα με πολύ μεγάλο μείγμα βιοκαυσίμων, άνω των 30%. Αυτά όμω τα καύσιμα είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό του συνόλου των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στι μεταφορέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δηλαδή και κάτω από το 1%. Okay. <clears throat> Uh, σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Σημειώνουμε τόσα μας είπατε και θα τα ξαναπούμε σίγουρα σε κάποια άλλη ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Έτσι ολοκληρώσαμε την εξέταση αυτού του σημείου. <clears throat> Ερχόμαστε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για τις επιπτώσεις στην υγεία της ισογλυκόζης. Έχουμε ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε την κυρία Αλεξάνδρα Νικολακοπούλου από την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ υγεία. Οπότε, παρακαλώ, Έχετε το λόγο για να μας παρουσιάσετε το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ που προσκαλέσατε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα της ισογλυκόζης. Θα σας ενημερώσω που βρισκόμαστε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σίγουρα μας ενδιαφέρει η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό το θέμα. Θέλω πρώτα απ' όλα να σας πω ότι πρόκειται για έναν όρο ο οποίος ε, αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και πρόκειται για ζάχαρη που παίρνουμε από δημητριακά και άμυλο. δεν είναι οι σουκρόζη που παίρνουμε από, το, από τα τεύτλα. Αυτό που επίσης είναι σημαντικό να καταλάβουμε εδώ είναι ότι η συνήθις ζάχαρη αποτελείται από γλυκόζη και φρουκτόζη, 50-50%. Και η ισογλυκόζη είναι μείγμα γλυκόζης και φρουκτόζης, αλλά με πολλές και διαφορετικές αναλογίες. Η όταν υπάρχει πολύ φρουκτόζη, 50% και 40% γλυκόζη, 42% φρουκτόζη και 53% γλυκόζη. Αυτές είναι οι παραλλαγές. Τώρα πώς χρησιμοποιείται η ισογλυκόζη. Αντικαθιστά, για παράδειγμα, τη ζάχαρη. η συνήθη τράπεζα που έχουμε από ζαχαρόταφλα ας πούμε. Υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα από τη χρήση της ισογλυκόζης. Είναι πιο φτηνή πρώτα απ' όλα, αλλά επίσης πρόκειται και για ένα ρευστό γλυκαντικό που έχει και άλλες ιδιότητες και χρησιμοποιείται συνήθως τα ποτά, σε μαρμελάδες και άλλα. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας εδώ ότι η ισογλυκόζη αποφεύγει την κρυστάλλωση και δεν κολλάνε τελικά οι ουσίες τις οποίες χρησιμοποιείται. Πρέπει συγχρόνως να έχουμε υπόψη μας ότι η κύρια ζάχαρη που χρησιμοποιείται μέχρι τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η κοινή ζάχαρη και υπήρχε έλεγχος στις αγωγές και την παραγωγή της ισογλυκόζης ελέγχεται από τις γεωργικές πολιτικές μέχρι τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό θα αλλάξει μετά από την τελευταία μεταρρύθμιση στην αγορά της αγοράς, η οποία ήταν πολύ ρυθμισμένη μέχρι τώρα, αλλά από φέτος και μετά δεν θα υπάρχουν ποσοστώσεις παραγωγής ούτε για τη σουκρόζη ούτε για την ισογλυκόζη, ούτε δηλαδή την κανονική ζάχαρη ούτε για την ισογλυκόζη. Αυτό θα οδηγήσει σε Αλλαγέ όσον αφορά την παραγωγή της ισογλυκόζης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι δύσκολο να προβλέψει κανεί το εύρο των αλλαγών αυτών. Κάποιοι στη Γενική Διεύθυνση Άγκρη πριν από λίγα χρόνια είπαν ότι μετά από τη μεταρρύθμιση αυτή θα πέσουν οι τιμές της ζάχαρης και η παραγωγή ζαχαρότευτλων θα αυξηθεί και η χρήση της ισογλυκόζης επίσης θα αυξηθεί πολύ πάνω από 12% ως γλυκαντικό. Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει ότι γίνεται η συζήτηση για το πώς θα αντιδράσουν οι σχετικές αγορές στην κατάργηση των ποσοστώσεων και συζητιούνται και οι επιπτώσεις στην υγεία με την επιπλέον χρήση της ισογλυκόζης. Θα πρέπει εδώ να πω επίσης ότι όταν κάναμε τη μεταρρύθμιση της αγοράς ε, ζάχαρης έγινε μελέτη αντικτύπου, αλλά δεν υπήρξε ειδικά για την υγεία μελέτη αντικτύπου. Σε επιστημονικό επίπεδο έχουμε ε, γνωμοδότηση από την ΕΦΣΑ, όχι ειδικά για την ισογλυκόζη, αλλά για την φρουκτόζη και γενικά για τις ζάχαρες. Όσον αφορά την ε, εφαρμογή και τους ισχυρισμούς όσον αφορά την υγεία, η ΕΦΣΑ σημειώνει στη γνωμοδότησή της ότι οι μεγάλες περιεκτικότητες σε φρουκτόζη μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις με δυσγλυπηδέμια, επιδεμία και άλλες ε, επιπτώσεις από την ε, συσσόρευση. Οι επιπτώσεις όμως αυτές σε χαμηλές δόσεις δεν παρατηρούνται. Και όταν μιλάμε για χαμηλές, εννοούμε 40 με 50 γραμμάρια την ημέρα. Η ΕΦΣΕ επίσης σημειώνει ότι οι αρνητικές αυτές επιπτώσεις της φρουκτόζης δημιουργούνται με κατανάλωση πάνω από 125 γραμμάρια την ημέρα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πολύ απίθανο να καταναλώσει κανείς όταν τρώει φυσιολογικά τόσο μεγάλες ποσότητες. Άλλη γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ έχει να κάνει γενικά με την κατανάλωση ζάχαρης. Και υπήρξε γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ για τις διαιτητικές τιμές από το 2010 για τους υδατάνθρακες και σύμφωνα με την γνωμοδότηση αυτή λέει η ΕΦΣΑ ότι δεν υπάρχουν αρκετές αποδείξεις για να αποφασίσει για ανώτατη επιτρεπτή τιμή κατανάλωσης ε, ζάχαρων. Πρέπει όμως εδώ να πούμε ότι πολλές χώρες μέλη έχουν εκδώσει συστάσεις για προσθετικά ζάχαρης που να μην είναι πάνω από 10% του, της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Και υπάρχουν και περιπτώσεις με 5 και 15%. Εδώ θέλω να αναφερθώ σύντομα στο θέμα της προστασίας των καταναλωτών για να εξηγήσω ότι η σογλυκόζη όταν χρησιμοποιείται στα τρόφιμα αναφέρεται στη σήμανσή τους ως ε, συστατικό. Και υπάρχει και ο κανόνας των ε, ενδεικτικών ε, σημάνσεων που επιτρέπει να αναφέρει κάποιος την περιεκτικότητα σε ισογλυκόζη επιπλέον αλλά συστατικά. Τώρα, άλλες δραστηριότητες. Θα υπάρξει αξιολόγηση στα πλαίσια ενό προγράμματος υγείας που μιλάει για τα επιστημονικά δεδομένα και την πολιτική που έχουμε όσον αφορά την κατανάλωση και τα ενεργικά στοιχεία τα οποία απορροφά ο οργανισμός μας και αυτό θα το έχουμε στα τέλη του 2017. Συγχρόνως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει και ρυθμιστικές και μη ρυθμιστικές πρωτοβουλίες όσον αφορά την κατανάλωση ζάχαρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, όπως γνωρίζουμε, από τον 13 Δεκεμβρίου του 2016 είναι η ενημέρωση όσον αφορά για το συνολικό ποσό ζάχαρων που περιλαμβάνεται στα τρόφιμα. Η δεδηλωμένη ποσότητα ε, ζάχαρης έχει να κάνει με τα μόνο ζαχαρόδια και δύο ζαχαρόδια που βρίσκονται στα τρόφιμα και έτσι συνοψίζεται η περιεκτικότητα γλυκόζης και φρουκτόζης, όπως και της ισογλυκόζης. Επίσης, η DG Santa στηρίζει τις εθνικές προσπάθειες για μη ρυθμιστικές πρωτοβουλίες και εδώ θα αναφέρω τη στρατηγική του 2007 για την Ευρώπη όσον αφορά την παχυσερκία σε σχέση με τα προβλήματα υγείας, που στηρίζεται από δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε συνεργασία με τις χώρες μέλη. Το Φεβρουάριο του 2011 η ομάδα υψηλού επίπεδου αποφάσισε ένα πλαίσιο για πρωτοβουλία σε θελοντική βάση όσον αφορά την περιεκτικότητα και το 2015 υπήρξε ένα παράρτημα το οποίο συμφωνήθηκε για την ε, πρόσθεση ζάχαρης που μιλάει για μείωση 10% της πρόσθεσης ζάχαρης μέχρι το 2010. Και υπάρχει και η πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις φυσικές δραστηριότητες και άλλες ε, δράσεις και εκεί αναφέρεται και επαναδιατύπωση της διατροφής. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχει υποχρέωση που έχει αναλάβει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι χώρες μέλη για τη μείωση της χρήσης της ζάχαρης στα τρόφιμα. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες πρέπει να ληφθούν υπόψη και όταν θα ετοιμάσουμε την, ε, και θα αξιολογήσουμε μάλλον την ε, μεταρρύθμιση της ε, ζάχαρης και την χρήση κυρίως της ισογλυκόζης. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε για τις εξηγήσει που μας δώσατε. Η κυρία Σαλτεμόζα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα όσα μας είπε. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα και πλούσιο στο περιεχόμενο. Αλλά είμαστε ειλικρινείς. Για μας τους σοσιαλιστές, και εδώ θα τα πω μα, έτσι, μας φαίνεται ανόητο να ε, προχωράμε σε αυτό το θέμα για την ισογλυκόζη στην υγρή μορφή, ενώ ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα με την υγεία, ότι δεν είναι ένα υγιεινό συστατικό. Εσείς λέτε ότι στα τέλη του 2017 θα έχουμε μία αξιολόγηση αντικτύπου. Τότε γιατί δεν περιμένουμε μέχρι τότε και τότε μόνο να ανοίξουμε την αγορά. Γιατί θέλουμε να την ανοίξουμε τώρα. Ας περιμένουμε τα επιστημονικά στοιχεία της μελέτης αυτής αντικτύπου. Γιατί δεν περιμένουμε. Λίγο, λίγοι μήνες μένουν μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Ας δούμε τότε κατά πόσο επιστήμονες μας λένε ότι όλα είναι εντάξει ή όχι. Ξέρω, θα πείτε ότι αν δεν γίνεται γιατί έχει ήδη ληφθεί απόφαση κτλ. κτλ. Έχουμε ήδη αποφασίσει να σταματήσουμε τις ποσοστώσεις, αλλά τώρα θα σας ρωτήσω αλλιώς. Ελέγχετε από κοντά τις επιπτώσεις στην υγεία από το άνοιγμα αυτό της αγοράς ζάχαρων τα επόμενα χρόνια. Προβλέπετε τέτοια παρακολούθηση από κοντά για τις επιπτώσεις στην υγεία, γιατί πρέπει να το ξέρουμε. Αν προχωράμε προς την λάθος κατεύθυνση, θα πρέπει να αντιδράσουμε. Επίσης, αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να υπάρχει χαμηλή απορρόφηση. Και τότε λέτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Όμως κοιτάξτε τι γίνεται στην Αμερικανική αγορά. Αυτό το σιρόπι, η ισογλυκόζη, χρησιμοποιείται κατά 50% σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα. Και δεν θα γίνει το ίδιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πιο φτηνό, όπως είπατε, και πιο εύχριστο ω συστατικό. Οπότε δεν θα γίνει το ίδιο και εδώ, όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τότε η απορρόφηση της ουσίας αυτής δεν είναι χαμηλή, θα αυξηθεί πάρα πολύ. Οπότε πρέπει να ξέρετε ότι οι σοσιαλιστές ανησυχούμε πάρα πολύ για τις επιπτώσεις στην υγεία αυτής της ουσίας. Αν μη τι άλλο, πρέπει να ελέγχουμε από κοντά την κατάσταση και να είμαστε έτοιμοι να δράσουμε να αλλάξουμε τακτική αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει επίπτωση στην υγεία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Γούγκετ. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή. Καταρχήν ε, για τις εξηγήσεις που μας έδωσε σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Εδώ αναφερόμαστε στις ε, επιπτώσεις της κατανάλωσης γλυκόζης στην υγεία ε, το ερώτημα είναι γιατί το κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Γιατί μας είπατε ότι ε, ο σχετικός ε, κανονισμός για την αγορά δεν θα ισχύει. Αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα ήταν ότι η εισαγωγή της ολοκληρικής μπορεί να περιορίζεται στο 50% του, του συνόλου της αγοράς της ζάχαρης. Δηλαδή 700.000 τόνοι ετησίω. Άρα λοιπόν αυτό που αναμένουμε μετά από την αλλαγή στα τέλη του έτους είναι ότι θα αυξηθεί αυτή η κατανάλωση θα τριπλασιαστεί δηλαδή έω ε, έως και 2,4 εκατομμύρια ε, τόνου. Ποιες ε, είναι ανησυχίες λοιπόν σε σχέση με αυτή την εξαιρετική αύξηση της κατανάλωσης. Να σας εξηγήσω. Έχουμε να κάνουμε με ένα βιομηχανικό ζάχαρο, το οποίο <clears throat> προέρχεται από άμυλο, συχνά ειδικότερα από άμυλο αργοσύντου. Άρα λοιπόν, λόγω της υγρής της μορφής, η ισογλυκόζη χρησιμοποιείται κυρίως στην ποτοπία, αλλά και στη ζαχαροπλαστική. Ε, οπότε έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα από οικονομική άποψη. Ισοπλικός. Είναι έως ε, ε, κατά 40% φθηνότερο. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν συζητάμε στην Επιτροπή ε, το ζήτημα αυτό. Κατά τη δική μου λοιπόν άποψη, η δεν είναι ε, υγιεινή, γιατί ε, μεταβολίζεται με διαφορετικό τρόπο από τον οργανισμό. Η φρουκτόζη, για παράδειγμα, μεταβολίζεται στο ε, σηκώτη και ε, τα όσα παράγονται από αυτή τη διαδικασία μπορεί να, ε, ε, αυξήσεις, να μειώσεις αύξηση της ινσουλίνης, πράγμα που μπορεί να έχει επιπτώσεις και στην παρουσίαση του διαβήτη. Ενώ κάποια πειράματα σε ορισμένα ζώα έχουν καταδείξει ότι υπάρχει αύξηση του λίπους στο σηκώδη. Ε, και αλλού έχει ε, βρεθεί αυτή η σύνδεση μεταξύ δηλαδή υψηλού λίπου στο σηκώδη και χρήση της γλυκόζης. Αφού λοιπόν ε, η υποτοπία και ζαχαροπλαστική θα αυξήσει προφανώς την χρήση αυτής της ισογλυκόζης, αυτό σημαίνει βέβαια ότι ειδικότερα τα παιδιά και οι νέοι που καταναλώνουν αυτά τα προϊόντα ενδεχομένω θα οδηγηθούν σε υψηλότερη παχυσαρκία. Στις ΗΠΑ η ισογλυκόζη χρησιμοποιείται ο Βρέο και φτάνει στο 50 Τη της συνολικής αγοράς ε, ζάχαρης και φοβούμαστε ότι θα έχουμε μια αντίστοιχη εξέλιξη και εδώ. Πέρα λοιπόν της παρακολούθησης, στην οποία μόλις αναφέρθηκε η συνάδελφος, ε, θα θέλαμε να ευαισθητοποιήσουμε ε, τους καταναλωτές μας και ιδιότερα τους νέους καταναλωτές μας ως προς το τι ακριβώς καταναλώνουν. Δηλαδή το γλυκό δεν είναι πάντοτε γλυκό και, το, και ζάχαρη δεν είναι πάντοτε ζάχαρη. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ε, ακριβή δεδομένα ως προς το πώς χρησιμοποιείται η ισογλυκόζη και χρειαζόμαστε και συγκεκριμένη σήμανση της ισογλυκόζης. Οπότε θα θέλαμε να ξέρουμε ποια είναι τα δικά σας σχέδια σε σχέση με αυτό ε, και νομίζω πως θα πρέπει να προβλέψουμε και συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τους ε, παραγωγούς. Δεν μπορούν δηλαδή, δεν θα, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ολογία περισσότερο ισογλυκόζη μόνο και μόνο για οικονομικούς σκοπούς. Δεν θα μπορούμε δηλαδή να, επιτρέψουμε να δοθεί προτεραιότητα σε οικονομικού ε, σκοπού, οι οποίοι θα επιτελούν τον ε, σκοπό τη προστασία τη υγεία των καταναλωτών μα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει ο κ. Πετιτσίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Επιτροπή που είναι παρούσα σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Εγώ θέλω να εστιάσω την προσοχή μου στις επιπτώσεις στην υγεία από την κατανάλωση σογλυκόζης. Γιατί όπως μόλι τώρα αναφέρθηκε υπάρχει ισογλυκόζη σε πολλά... Ε, αναψυκτικά τα οποία τα καταναλώνουν κυρίως οι νέοι και στα γιαούρτια και σε πολλά άλλα γλυκά αυτά που τα καταναλώνουν κυρίως τα παιδιά η Κομισιόν μίλησε επίσης για τη λειτουργία της ισογλυκόζης είναι ένα συστατικό ε, το οποίο επιτρέπει να μην κολλάνε τα συστατικά ενός γλυκού μεταξύ τους. Σα ε, σας είπα επίσης ότι κύριος αποδέκτης είναι τα παιδιά θα πρέπει να εξετάσουμε και άλλα στοιχεία, όπως όχι μόνο την παχυσαρκία, και, την, και το διαβήτη, γιατί ο ισογλυκόζη ε, συνδέεται και με πολλές άλλες ε, βιομηχανικές ζάχαρες. Να έχουμε κατά νου ότι όλα αυτά ε, μας ανησυχούν, παρουσιάζεται σημαντική αύξηση αυτών των ασθενειών και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να εξετάσουμε τις πηγές της κάθε αυτής ασθένειας. Εγώ συμφωνώ με αυτά που είπε η συνάδελφος κυρία Σαλντεμός, δηλαδή να περιμένουμε τη μελέτη αντικτύπου πριν ανοίξουμε την αγορά σε αυτή την ουσία και πρέπει επίσης να προβάλλουμε την ε, διαπαιδαγώγηση σε θέματα διατροφής γιατί η ενημέρωση σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν και σωστές ετικέτες, σωστή σήμανση και ερωτώ την Κομισιόν. Ε, η παρουσία της ισογλυκόζης είναι υποχρεωτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει, μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο σιρόπι γλυκό και στην ισογλυκόζη. Η κυρία Ντάλη. Um, Ευχαριστώ. Ε, πρόεδρε, συμμερίζομαι τις ανησυχίες όλων των συναδέλφων και θα σα εξηγήσω γιατί. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στο σύνολό της, αλλά και τα κράτη-μέλη, επανειλημμένα ε, εδώ και κάποια χρόνια προσπαθούν να μεώσουν την παχυσαρκία αλλά και τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με το διαβήτη που είναι βέβαια ένα πρόβλημα υγείας αλλά και οικονομικό πρόβλημα ε, για τα επιμέρους κράτη-μέλη και για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δυστυχώς ε, πολλές φορές όταν αρχίσουμε να κάνουμε λόγο ε, για χρήματα αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε τις διαστάσεις του προβλήματος. Οπότε θα πρέπει να το κάνω και εγώ αυτό. Εγώ προέρχομαι λοιπόν από τη Μάλτα, από ένα νησί της ε, Μεσογείου, όπου δυστυχώς και η παχυσαρκία και ο διαβήτης είναι ιδιαίτερα εκτεταμένα προβλήματα υγείας. Είναι δηλαδή ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι μας. Αν, σας αν μου επιτρέπετε να σας δώσω κάποια στοιχεία, να σας πω ότι η πλειοψηφία των ατόμων που πάσχουν από διαβήτη πάσχουν και από παχυσαρκία. Ε, και παχυσαρκία και ο διαβήτης τύπου 2 κοστίζουν 53 εκατομμύρια ευρώ στη Μάλτα, που αντιστοιχεί στο 5% του συνόλου της δαπάνη υγείας ε, στη, Μάλτα. Εάν δούμε ε, την κατάσταση στα 28 κράτη-μέλη, είναι ακόμα πιο ανησυχητική η κατάσταση σε ό,τι αφορά την παχυσαρκία. Ε, πάνω από το ίμιση των ενηλίκων του ενήλικου πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρβαρη ή είναι υψηλότερη από τον τεκνόμενο βάρο. Και σε ό,τι αφορά το κόστο, 81 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το κόστος της βαχυσαρκίας ενώ το κόστος του διαβήτη 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Και σε ορισμένα κράτη-μέλη ε, αυτά τα ποσοστά ή αυτά τα νούμερα αντιστοιχούν στο 10% του συνόλου του προπολογισμού για την υγεία. Οπότε ας δούμε τα πράγματα, ας τα βάλουμε στη σωστή προοπτική. με αυτά τα χρήματα τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να επενδύσουν ε, ε, σε πολλούς άλλους τομείς όπου θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών τους. Οπότε πραγματικά ανησυχώ, ανησυχώ σοβαρά και για, μας, για μένα προσωπικά είναι απαράδεκτο ε, να λέμε ότι δεν γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος της ε, κατάργησης αυτής της ε, ποσόστοσης σε ό,τι αφορά τη ζάχαρη. Γιατί ακριβώ χάρη σε αυτή την ποσόστοση έχουμε επιτρέψει το να μην υπερβαίνει το 5% των συνολικών εισαγωγών ή ισογλυκόζη. Αλλά από αυτό που αντιλαμβανόμαστε μέσα στα 6 χρόνια αυτό το ποσοστό θα τριπλασιαστεί. Άρα λοιπόν δεν είναι αστείο εδώ. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Και αν δούμε τις μελέτες σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις της ισογλυκόζης στην υγεία είναι σοβαρές. Βλέπουμε δηλαδή ότι έχουμε να κάνουμε διαβήτη τύπου 2, έχουμε να κάνουμε παχιασαρκία, δηλαδή ζητήματα που θα επηρεάσουν την ποιότητα ποιότητα ζωή όχι μόνο των ενηλίκων μα, αλλά και των ε, νεότερων γενιών μας, πράγμα που με ανησυχεί ακόμα περισσότερο. Σε κάποια φάση αναφερθήκατε στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων. Έγινε μια δήλωση από την ΕΦΣΑ όπου ανέφερε ότι μελέτες οι οποίες ε, συνέκριναν ε, την ε, κατανάλωση αναψυκτικών που περιέχουν φρουκτόζη, ζάχαρη ή γλυκόζη διαπίστωσαν ότι όπου υπάρχει υψηλή περιοκτικότητα σε γλυκόζη εμφανίζουν περισσότερο ζάχαρα στο αίμα, υψηλότερη συσσόρευση λιπανόλου στο σηκώτη που μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακά προβλήματα και ούτω καθεξής. Δηλαδή μιλάμε για σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και εδώ κάνω λόγο για μια μελέτη της ΕΦΣΑ του 2013 και τώρα έχει γίνει αξίωση από την πλευρά των κρατών μελών για περαιτέρω ε, μελέτη, οπότε θα ήθελα να μου πείτε ποια ήταν τα πορίσματα της ελόγω ε, μελέτης, προκειμένου να αντλήσουμε κι εμείς κάποια διδάγματα. Έχει ε, σχεδιάσει η Επιτροπή κάτι έτσι ώστε να διασφαλιστεί το ότι ε, τα αναψυκτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον δεν θα περιέχουν τόσο υψηλό ε, ποσοστό φρουκτόζης. Ε, και από εκεί και μετά σε ό,τι αφορά τη σήμανση σε σχέση με τα GMOs, τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Τα ένζημα δηλαδή συνήθω που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή της δεν είναι υποχρεωτικό να αναφέρονται και ούτε υπάρχουν σχετικές υποχρεώσεις σε επίπεδο έτη και το στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω νομίζω πως οι καταναλωτές μας οφείλουν να γνωρίζουν πάντοτε τι καταναλώνουν, τι τρώνε και τι πίνουν, οπότε θα πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώ εάν θα καταργηθούν οι ε, περιορισμοί σε ό,τι αφορά την ισογλυκόζη, τι περιλαμβάνει αυτή η ισογλυκόζη. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ζάχαρη είναι ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα που γλυκαίνουν τα πράγματα, αλλά με την ε, ζάχαρη προκύπτουν και προβλήματα στην υγεία. Προκύπτει παχυσαρκία, ε, σαπίζουν τα δόντια, διαβήτης, υπέρταση και πολλές άλλες ασθένειες. Η σογλυκόζη είναι ένα υποκατάστατο της ζάχαρης και η κατανάλωσή της αυξάνεται. Και αυτό που είναι σίγουρο ότι πρόκειται για βιομηχανική ζάχαρη, η οποία είναι και σχετικά φτηνή. Ε, υπάρχουν, ε, υπάρχει μια ποσόστοση σχετικά με την ισογλυκόζη, αλλά αν καταργηθεί η ποσόστοση θα αυξηθεί και η κατανάλωσή της. Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε ότι η ζάχαρη αυτή, το υποκατάστατο ζάχαρης, ε, μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην υγεία. Και επιστημονικές μελέτες έχουν καταδείξει ότι η χρήση ισογλυκόζης στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, σημαίνει αν πίνει κανείς ε, ένα ποτήρι οτιδήποτε την ημέρα κενόμενο από ισογλυκόζη Αυτό ικανοποιεί τις ανάγκες του ατόμου σε ζάχαρη για ολόκληρη την ημέρα. Ο διαβήτης είναι ένα μεγάλο πρόβλημα κατά τον 21ο αιώνα. Ο διαβήτης τύπου 2 που εμφανίζεται σε άτομα που χρησιμοποιούν ισογλυκόζη Ο διαβήτης αυτός σε άτομα νεαρής ηλικίας Λοιπόν, ο διαβήτης αυτός εμφανίζεται κυρίως σε, άτομα νεαρής ηλικίας τα οποία είναι ινσουλινοεξαρτώμενα και στην περίπτωση αυτή η ισογλυκόζη είναι επικίνδυνη. Σε γενικές γραμμές η ισογλυκόζη κρίνεται ασφαλής, ε, αλλά θα πρέπει να έχουμε κατά νου και ότι δεν πρέπει να γίνεται υπερβολική κατανάλωση ισογλυκόζης. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή μήπως έχει κατά νου κάποιες εκθέσεις ε, σχετικά με τη χρήση υποκατάστατων της ε, ζάχαρης και επίσης θα ήθελα να γνωρίζω ποιες θα ήταν και επιπτώσεις αν ήταν ελεύθερη η χρήση ισογλυκόζης, χωρίς περιορισμούς. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, αλλά η ίδια η βιομηχανία μπορεί να περιορίσει τη χρήση της ισογλυκόζης. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι συνέπειες από τη χρήση της ισογλυκόζης μπορεί να είναι δραματικές και εγώ νομίζω ότι πρέπει απαραίτητα να, συνθέσουμε, να συντάξουμε μια έκθεση για τις επιπτώσεις της ισογλυκόζης στη δημόσια υγεία, στους, στην υγεία των Ευρωπαίων. Ευχαριστώ, κύριε Κάντμπαχ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την έκθεση και νομίζω ότι αυτά που λέξανε εδώ κατέδειξαν με απόλυτη σαφήνεια ότι φοβόμαστε πως αυτή η απόφαση Κομισιόν ακολουθεί λάθος κατεύθυνση. Εγώ ε, θα σας αναφέρω μία έκθεση ε, όπου ο κύριος Ροζάριο, εκπρόσωπος της Επιτροπής Γεωργίας, ε, ρωτήθηκε τελικά ε, Πώς προέκυψε αυτή η απόφαση και είπε και παραθέτω είναι μια απόφαση όπου η γεωργική πολιτική ακολουθεί την κατεύθυνση γενικότερα που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος της παράθεσης. Μάλλον όχι, συνεχίσε και λέει δεν είναι πολιτική για τους καταναλωτές ούτε πολιτική υγείας. Αυτά είναι τελείως διαφορετικά θέματα. Τέλος παράθεση και ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός της NDF είπε τότε στο συμπέρασμα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ακολουθείται γεωργική πολιτική χωρίς να λαμβάνεται καν υπόψη να λαμβάνουν υπόψη τα θέματα της υγείας. Αν δούμε όμως το άρθρο 168 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί αναφέρεται με απόλυτη σαφήνεια ότι όταν χαράσσονται ενωσιακές πολιτικές, πρέπει να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας υγείας. Άρα δηλαδή και μόνο να ακούσει κανείς το τι ελέγχεται εδώ σήμερα. Δεν χρειάζεται καν να έχει ενδελεχή μελέτη και μόνο από αυτά τα σημερινά καταλήγουμε στο ότι υπάρχει παραβίαση του άρθρου 168, διότι η προστασία της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών σαφώς ε, θεωρείται κατώτερη του ανοίγματο της αγοράς ε, και εγώ ε, δεν καταλαβαίνω το άνοιγμα αυτό της αγοράς ποιον Ευρωπαίο θα ωφελήσει θα ήθελα να εξετάσουμε το εξή. Μήπω έχουμε μια κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μια απόφαση που σαφέστατα και παραβιάζει τι ευρωπαϊκές συνθήκε. Ευχαριστούμε. άλλο παρακαλώ. Από ό,τι βλέπω κανένας δεν θέλει το λόγο. Επανέρχομαι λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ακούσουμε τη δική της την άποψη. Σας ευχαριστώ. Ακούσαμε προσεκτικά τα σχόλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως είπε και η κυρία Σάλντε Μόζε, δεν μπορούμε να περιμένουμε τώρα ότι θα λάβει χώρα η μεταρρύθμιση για τα ζάχαρα και πρέπει να περιμένουμε την ε, μελέτη αντικτύπου για την ισογλυκόζη πρώτα. Αυτό που είπα εγώ για την ε, συνολική αναθεώρηση δεν είναι αξιολόγηση αντικτύπου αυτή καθεαυτή. Πρόκειται για την, ε, τόσα έχουν γραφτεί και τόσα γνωρίζουμε όσον αφορά την, επιπτώσεις από τη χρήση της γλυκόζης και της ογλυκόζης. Αυτό που είναι ενδιαφέρον βέβαια να σημειώσουμε είναι ότι η ΕΦΣΑ μετά από αίτημα σκανδιναβικών χωρών, Νορβηγίας, Σουηδίας, Δανίας, Φιλανδίας και Ισλανδίας, εξετάζει και έχει δεχτεί εντολή για επιστημονική γνωμοδότηση όσον αφορά τις ποσότητες της ημερήσιες απορρόφησης και για τους κινδύνους από την απορρόφηση ζαχάρων από όλες τις πηγές. Σουκρόζη, φρουκτόζη, γλυκόζη, ε, υδροπτικό άμυλα, φρουκτόζη και άλλα παρασκευάσματα ζαχάρων που προστίθενται στα τρόφιμα κατά την παρασκευή τους. Όπως καταλαβαίνετε το χείρημα αυτό θα κρατήσει αρκετά. Η ΕΦΣΑ θα συναντηθεί με όλους τους ενδιαφερόμενους βάσει της διαδικασίας ε, διαβούλευσης και θα έχει και δύο επίσημες διαβουλεύσεις το πρώτο ήμιση του 2018 με τον κόσμο και θα έχουμε γνωμοδότηση στα τέλη του 2019. Αυτό που βλέπουμε δηλαδή και με την ΕΦΣΑ ότι υπάρχει δυνατότητα να ενισχυθεί περισσότερο αυτό το εγχείρημα με την πτυχή που έχει να κάνει με τις επιπτώσεις στην υγεία της ισογλυκόζης. Όμως θέλω να επενθυμίσω ότι αυτά που είπε η κυρία Ντάλη για την γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ που αναφέρεται σε αρνητικές επιπτώσεις πρόκειται για αρνητικές επιπτώσεις εφόσον υπάρχουν υψηλά επίπεδα απορρόφησης, φρουκτόζης. Γιατί αυτό είναι συνήθως, είτε πρόκειται για την κοινή ζάχαρη είτε για την ισοκλικόζη. Μιλάμε και 125 γραμμάρια την ημέρα απορρόφηση. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ. Είναι απίθανο να καταναλώσει κανείς όταν τρώει φυσιολογικά τέτοιες ποσότητες. Η ιδέα τώρα του ελέγχου που είπατε. Να παρακολουθήσουμε τις επιπτώσεις από την κατανάλωση ισογλυκόζης. Είναι ενδιαφέρον ως ιδέα. Εμείς δεν μπορούμε να δεσμευτούμε τώρα ότι θα γίνει, αλλά αυτό που θα μεταφέρουμε θα το βάλουμε στην ημερήσια διάταξη για να το συζητήσουμε με τις χώρες μέλη και με τους ενδιαφερόμενους, αυτό τον δεχόμενο δηλαδή παρακολούθησης. Ρωτήσατε και για την σήμανση, για τις ετικέτες. Ναι, όπως σας είπα και πριν, η ισογλυκόζη πρέπει να αναφέρεται στα συστατικά, στη σήμανση, αλλά η ισογλυκόζη είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στην γεωργική νομοθεσία μας. Αυτό που συνήθως βλέπουμε στα συστατικά είναι γλυκόζι, φρουκτόζι, σιρόπι, κάτι δηλαδή που έχει να κάνει με σιρόπι από γλυκόζι και φρουκτόζι ανάλογα ε, με τη μία με την άλλη σειρά, ανάλογα με το πιο κυριαρχεί στα συστατικά. Και επιπλέον έχουμε και τη θρεπτική αξία που βέβαια αυτή αναφέρεται για όλα τα ζάχαρα και όχι ειδικά για την ισογλυκόζη. Αυτά νομίζω μπορώ να απαντήσω. Πάντως, σημειώνουμε τις ανησυχίες σας και θα εξεταστούν παρετέρω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα συζητηθούν με τις χώρες μέλη και του ενδιαφερόμενους στα διάφορα φόρα όπου συζητείται το θέμα αυτό της υγείας στη διατροφή. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Έτσι ολοκληρώνεται η συνεδρίασή μας. Στις 2 το απόγευμα πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή πάλι και το Ελεκτικό Συνέδριο για την ανεξαρτησία και την σύγκρουση συμφερόντων. Δύο η ώρα λοιπόν, εδώ θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ.